Colegas, vamos a proceder a las explicaciones de Έχουμε 16 συναδέφους που επιθυμούν να, εκφράσουν μια επεξήγηση ψήφου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι η διαδικασία επιτρέπει να υποβάλουν γραπτό στο κείμενό τους έτσι δεν πρέπει λοιπόν να βιαστούν να κάνουν γρήγορα την παρέμβασή τους και το αντίθετο κιόλας ε, θα διαβιβαστεί στην εφημερίδα των πρακτικών ε, με μεγαλύτερη ακρίβεια έτσι η παρέμβασή τους. Έχουμε επεξηγήσει ψήφου για την συμφωνία πλαίσιο για την, την Ευρωβουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθένας θα έχει δύο λεπτά από τους αγορητές και πρώτος ένα λεπτό, ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρο. Πρώτο θα λάβει τον λόγο ο κύριο Κλεμέντε Μαστέλα. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Μαστέλα. Δεν παρίσταται ο κύριος Μαστέλα. Δεν είναι παρόν στην αίθουσα. Έτσι λοιπόν θα λάβει τον λόγο για ένα λεπτό. Ναι, κύριε Μαστέλα, έχετε τον λόγο λοιπόν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να με. Τι δεν με ακούτε. Α, μ' ακούτε. Ευχαριστώ. Η συμφωνία πλαίσιο που μόλις ψηφίσαμε βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό. Πρόεδρε, δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούγομαι. Όχι, ακούγεστε, ακούγεστε. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα της ώρας. Toma usted la palabra, señor Mastella. Migliora considerevolmente il ruolo del Parlamento europeo Βελτιώνει λοιπόν την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα ρόλο ο οποίο έχει ούτω ή άλλω ενδυναμωθεί με την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δώσαμε την εμπιστοσύνη μα στον κύριο Μπαρόζο και περιμένουμε τώρα από πλευρά του την ανταπόκρισή του σε σχέση με τι μεγαλύτερε μα προτεραιότητε. Θεωρούμε σημαντική μια πιο στενή συνεργασία ώστε να έχουμε τακτικό διάλογο ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα ενημέρωση και τακτικό διάλογο, όπως είπα, στις ε, βασικές, στα, θέματα και στις βασικές νομοθετικές προτάσεις. Τα θεσμικά μας όργανα θα κληθούν, κύριε Πρόεδρε, να υλοποιήσουν την δημοκρατική μέθοδο, όπως αποκαλείται, μέσω της υλοποίησης ε, μια ειδική εταιρική σχέσης με στόχο να καθοριστεί ο ευρωπαϊκός έλεγχος στα διάφορα επίπεδα. Μεγαλύτερη ευθύνη για την Κομισιόν αλλά και για μας που είμαστε οι άμεσοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι στόχοι κύριε Πρόεδρε και κλείνω απαιτούν ε, Μεγάλη αφοσίωση από πλευρά ε, Κοινοβουλίου, Κομισιών, Συμβουλίου, Κυβερνήσεων, Εθνικών Κοινοβουλίων για να μπορέσουμε να, να εγγυηθούμε την πορεία τη Ευρώπη για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σα ευχαριστώ, κύριο Πόσελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι και υπέρ της Συμφωνίας Πλαισίου που είναι μια ιστορική πρόοδος ως αποτέλεσμα. Γιατί καταψήφισα τώρα παρόλα αυτά το ψήφισμα επειδή εχθές το οποίο ε, υπευλήθη ως έτοιμο κείμενο δεν μπορέσαμε, δεν μπόρεσα να την εξετάσω σε βάθος και οι λεπτομέρειες, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και υπάρχουν και επιφυλάξεις για κάποιες διατυπώσεις όσον αφορά για παράδειγμα τα δικαιώματα επιμέρους ε, βουλευτών ή τον κίνδυνο να υπάρξει εδώ κάποια κρυφή ας το πω έτσι συμφωνία όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρίσκεται στη διάσκεψη των πρόεδρων. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρξουν κάποιες διορθώσεις στο κείμενο και δίκαια αναφέρθηκε ότι έχει περισσότερε εξουσίε τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάζεται στενή συνεργασία και σχέση συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν χρειάζεται λιγότερη, αλλά περισσότερη δημοκρατία και δημοκρατικά δικαιώματα. Μεγαλύτερη δημοκρατία λοιπόν και στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό καταψήφισα αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντανίερ Χαμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο ημικύκλιο δεν μπορεί κανείς να πιστεύει ότι οι 27 αυτοί υποψήφοι είναι καταλληλότεροι ως επίτροπη από τους 500 εκατομμύρια πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρώπης και έχει την πρωτοβουλία για την νομοθετική πράξη, για το νομοθετικό έργο. Ποιο όμως της προσδίδει αυτή την εξουσία. Μια σειρά από υποψηφίους που προκύπτουν από συμβασμούς, από ε, διαδικασίες ε, δούνε και λαβήν με τις εθνικές κυβερνήσεις ή ως ε, ανταπόδοση για υπηρεσίες. Για να μιλήσω λοιπόν για την υποψήφια της δική μου τη Βαρόνη Άστον. Η γαλλική κυβέρνηση την καταδικάζει γιατί δεν μιλάει τα γαλλικά. Υποτευτεί, μα κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το λιγότερο από τα μειονεκτήματά της. Η Βαρόνη Άστον δεν έκανε τον κόπο ποτέ να εκτεθεί στην ε, καθολική ψηφοφορία. Πώς λοιπόν μπορεί να δώσει η Ευρώπη στο Ιράν την Κούβα διδάγματα για τη δημοκρατία όταν η υπεύθυνη για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρώπης η ίδια δεν έχει εκλεγεί άμεσα. Η κυρία και οι φεντεραλιστές φίλοι της μας, μας κατηγορούν ως αντιευρωπαϊστές. Όταν ε, έγινε ο αγώνας όμως για τα πυρηνικά εάν είχαν κερδίσει στις ε, διαδηλώσεις τους και είχαν επιβάλει τις νόμες τους, θα ήταν ακόμα διχασμένη η Ευρώπη, θα είχαμε ακόμη ψυχρό πόλεμο. Ο Πρόεδρος διακόπτη. Ξεπεράσατε το χρόνο σας. Τώρα θα λάβει τον λόγο, θα έχουμε επεξηγήσει ψήφου τώρα όσον αφορά την παρουσίαση του Σώματος των Επιτρόπων. Πρώτος θα λάβει τον λόγο ο κύριος Ουσπάσνικ, παρακαλώ. Ατσού. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τη νέα Επιτροπή, τον Συλλογικό Όργανο. Επισημάνοντας όμως κάποια δικαιογονότα που λησμονήθηκαν και στη συζήτηση δεν αναφέρθηκαν ούτε από τις πολιτικές ομάδες, από τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων, ούτε στην Ολομέλεια υπεγράμμισα την ε, διαδικασία που επελέγει για το διορισμό και τους υποψηφίους. Και είχα πει, ομιλώντας εκ μέρους της ε, ομάδας μου, ότι θα πρέπει τους υποψηφίους να τους ε, υποστηρίξουν προκαταβολικά τα δύο τρίτα των εθνικών τους κοινοβουλίων και μετά να προχωρήσουν από τι εθνικέ κυβερνήσει υποψηφιότητε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι μια πρόταση που είχα κάνει. Και επίση μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι η νέα Επιτροπή θα πρέπει ιδιαίτερα να διαφυλάξει τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει έναντι εισαγωγών από χώρες οι οποίες δεν υιοθετούν αρχές αντίστοιχες με τις δικές μας όπως την περιβαλλοντική προστασία της κοινωνικής εγγύηση και τους δημοκρατικούς θεσμού αυτά θα πρέπει να αναγνωριστούν ως όρια εκτερών ουκάνευ για να ε, ε, εγκριθεί η εισαγωγή προϊόντων από τέτοιες χώρες. Γιατί από τέτοιες χώρες θα γίνονται εισαγωγές ε, ε τίθεται σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Ο κύριος Χάναν έχει τον λόγο για άλλη μια φορά και έτσι μπορεί να συνεχίσει την προηγούμενη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να πού βρισκόμαστε. Η Βαρόνη Άστον και οι φεντεραλιστές ε, φίλοι της μας ε, κατηγορούν ως αντιευρωπαϊστές, αλλά εάν είχαν κερδίσει την εκστρατεία τους κατά πυρηνικών θα είχε παραμείνει διχασμένη η πυρός μας και εκατοντάδες εκατομμυρίων πολιτών θα ε, βρίσκονταν ακόμα εκτεθειμένοι στην μαξιστική τυραννία. Κανένας πραγματικός Ευρωπαίος, κανένας πραγματικός δημοκράτης δεν μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια υποψήφια. Εκφράζοντα λοιπόν θετική ψήφο μόνο και μόνο γιατί αυτοί έχουν ε, τοποθετηθεί υπέρ της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρου, ουσιαστικά mm. καταδικάζει το κοινοβούλιο των εαυτών του. Πολύ καλά συνάδελφε. Τώρα θα περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου όσον αφορά τον διορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα η κυρία Ιβαζανίκη παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη που υπερψήφισα αυτό το νέο σύνολο επιτρόπων. Είμαι ικανοποιημένη γιατί είδα άνδρες και γυναίκες πολύ προετοιμασμένους με ξεκάθαρα και συγκεκριμένα προγράμματα. Εύχομαι καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, καλή δουλειά στον Αντώνιο Ταγιάννη γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύτιμος που μπορεί να συμβάλλει ε, στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Και έπειτα, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης θα πρέπει να υπογραμμίσω την εξαιρετική εντύπωση που αποκόμισα από την κυρία Γεωργίευα. Μια γυναίκα πραγματικά αποφασιστημένη και ικανή. Θα είναι μεγάλη ε, χαρά για την Επιτροπή Ανάπτυξη να συνεργαστεί μαζί τη. Εύχομαι καλή δουλειά σε όλου. Σα ευχαριστούμε κυρία Ζανίκη. Και τώρα... Σα ευχαριστώ κυρία Ζανίκη. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριο Ζιά, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είναι σημαντικό να χαιρετήσουμε το ότι θα έχουμε μια αποτελεσματική δραστήρια Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, μια ισότιμη συνεργασία μεταξύ Ευρωβουλή και Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασιστική σημασία αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Η σημερινή αυτή συμφωνία αποτελεί τα βάθρα αυτή τη συνεργασία. Θα έχει απόλυτε εξουσίε απόφαση η Ευρωβουλή και θα είναι ισότιμη έναντι τη Επιτροπή και αποφάσεων που θα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Υπό αυτό το πνεύμα θα συνεργαστούμε σε βάθο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με εμπιστοσύνη από πλευρά μα, αλλά όχι χωρί επικριτικό πνεύμα και κριτικό πνεύμα. Αυτό δείχνει ότι τίποτα δεν θα μπορεί να παρακάμπτει το Κοινοβούλιο ως απόφαση. Και θα ήθελα να μπορέσουμε και για τα θέματα SWIFT να μπορεί το Κοινοβούλιο να αρθρώσει λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Αντωνιώτση, παρακαλώ. Presidente, colleghi, ho votato a favore della Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Υπερψήφισα την Επιτροπή Παρόζου γιατί είμαι βέβαιος πως θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις που μας ε, ε, που μας, που μας υποχρεώνει η οικονομική κρίση να τις ε, αντιμετωπίσουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα. Επίσης, ε, για ορισμένα θέματα τα οποία μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή, θα ήθελα να αντιμετωπιστούν με την δέουσα προσοχή. Ας πούμε, οι περιφερειακές πολιτικές που έχουν σημαντικό ρόλο όταν μιλάμε για ανάπτυξη και των περιφερειών μας και που δεν θα πρέπει να παραμένουν στα ψίχουλα που παίρνουν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ε, πολύ συχνά μεγάλη ενεργία πλήττει τα αστικά κέντρα και θα ήθελα ειδικά ε, μέσα ε, να δοθούν και να ξαναμπούν στις προτεραιότητες για την πολιτική στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εύχομαι καλή δουλειά στην καινούρια Επιτροπή. Σας ευχαριστώ και ο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 Σας ευχαριστούμε, κύριος Higgins, παρακαλώ. Eh, Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα τον διορισμό της νέας επιτροπής γιατί στην ουσία πρόκειται για την συνέχιση της νέας νεοφιλελεύθερης δεξιάς πολιτικής που κατέληξε στην καταστροφή των οικονομιών πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Αυτή υποτιθέμενη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχτεί πως είναι το ίδιο παλιό κρασί που έχει όμως γίνει ξύδι με τις ίδιες πολιτικές θα έχει αυτό καταστροφικές συνέπειε για τις ζωές ε, των ε, ανθρώπων τη εργατική τάξη με μαζική ανεργία και μείωση του επίπεδου ζωής. Οι κρίσει που ζοβούν στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία είναι ε, παραδείγματα ή και μάλιστα η Επιτροπή συμφωνεί πως η εργατική τάξη είναι αυτή που θα πληρώσει την ύφη ενώ οι τράπεζε είναι αυτέ που παίρνουν τα λεφτά μόλι χτυπηθούν από την κρίση θα θέλαμε να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή, δημοκρατική και σοσιαλιστική ε, Ευρώπη και αυτό σημαίνει καταψήφιση αυτής της νέας Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ξαναπάρτε τον λόγο για μια τρίτη επεξήγηση. Κύριε Χάναν, παρακαλώ. Παρατούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που αποσύρατε το αίτημα και έτσι εξοικονομούμε χρόνο. Ο κύριος Σανέκερ, παρακαλώ. Eh, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σε πολλές παρεμβάσεις από αυτές που ακούσαμε στο σώμα, δηλαδή που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την απόρριψή της, μπορεί κανείς ε, ένα συμπέρασμα να συναγάγει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει απλά την πορεία της και την Ισλαμική Τουρκία θα, τις, θα την αφήσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων λένε ότι εμείς θα θέλαμε να αποφασίσουμε αυτό το θέμα με δική μας ετοιμιγορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την προσπάθειά της εκατομμύρια και θα έλεγα και θα τολμούσα να πω δεκάδες εκατομμύρια ανέργων να μπορούν να ε, συνεχίζουν ως μετανάστες να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρότι κανένας από τους νέους επιτρόπους δεν είναι πρόθυμος να κάνει οτιδήποτε. Και αυτοί είναι αρκετοί λόγοι να καταψηφίσει κανείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ συνάδελφε λέγει ο Πρόεδρος. Τώρα ο κύριος Σπερώνη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Για τη νέα αυτή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε συγκεκριμένες και επαρκείς απαντήσεις που να δόθηκαν στα ερωτήματα και στα θέματα όπως παράδειγμα παράνομη μετανάστευση όσον αφορά την ίδια την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν αρκετός λόγος, επαρκής λόγος για να πούμε όχι κύριοι, απορρίπτουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν εγκρίνουμε αυτό το πρόγραμμα. Όμω υπάρχουν και άλλοι παράγοντες και στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως ο πρόεδρός της τι έκαναν τις ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτής της Ευρωβουλής ε, δεν ε, θέλησαν να, να τις πάρουν στα σοβαρά. Αυτό θα ήταν κάτι σαν, ας το πω έτσι, κατά της δημοκρατίας. Εμείς οι ίδιοι είμαστε οι εκπρόσωποι, αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών μας. Αν το δικαίωμα πρωτοβουλίας το δικό μας δεν είναι σεβαστό λοιπόν και οι δικές μας προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και για το άρθρο 125 της συνθήκης που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Σκαμάν, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εξετάζοντας τα πρόσωπα των υποψηφίων σήμερα, πιστεύω θα μπορούσαν όλοι οι συναδελφοί να συμφωνήσουν ότι κάποιοι ήταν καλοί, κάποιοι πολύ καλοί, κάποιοι κακοί και κάποιοι πραγματικά ανεπαρκείς. Δυστυχώ όμως κάποιοι δεν έδωσαν απαντήσει για το παρελθόν τους. Εμείς όμως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε επιμέρους επιτρόπους και έτσι ε, είχαμε μία επιλογή. Ή να τους εγκρίνουμε όλους στι θέση, στις θέσεις τους ή να τους απορρίψουμε όλους. Λυπηρή επιλογή και γι' αυτό προτίμησα να απόσχω τη ψηφοφορία. Ο κύριος Μπαρόσο μίλησε για ανταπόκριση στην κρίση. Εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε στην κρίση, καλό θα είναι να μην συσσωρεύουμε το ένα νομοθέτημα μετά το άλλο, αλλά να κάνουμε πρώτα απ' όλα αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητα των οδηγιών, όπω οι παραδείγματα για τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ταμείων και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που έχει σαν αποτέλεσμα να καταπνίξει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, να διώξει το χρήμα από την Ευρώπη και να το μεταφέρει σε άλλε χώρε. Εάν αυτό μόνο κοιτάγαμε, θα είχαμε κάνει μεγάλο ε, πολλά για την Ευρώπη. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Δέβα έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Ο κύριος Δέβα χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εμένα με εκλέγουν οι ψηφοφόροι μου στην Νοτιοανατολική Αγγλία για να ψηφίσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεταρρυθμίσεις και όχι για τα τρέχοντα και τετριμένα, για τα ίδια αυτά που μας παρουσιάζει ως ιδέες. Ναι, ο κύριος Παρόσο έχει την προσωπική μου εμπιστοσύνη, όπως και κάποιοι άλλοι από τους επιτρόπους, τους οποίους έχω στο παρελθόν γνωρίσει και έχω έρθει σε επαφή μαζί Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να εγκρίνω ολόκληρη την Επιτροπή ω συλλογικό όργανο, γιατί ο κάθε επίτροπο είναι μοναδικός, έχει στην πολιτική του ιστορία και κανένας δεν μπορεί στην δημοκρατία να έχει εξουσία όπως αυτή που έχει τώρα η Επιτροπή μας, δηλαδή την εξουσία για νομοθέτημα, για ε, εκτελεστική εξουσία και πάλι χωρίς ε, έλεγχο δημοκρατικό και χωρίς επιμέρους εκλογή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό ο κύριος Κλάις, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταψήφισα τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπορεί κανείς να πει η νέα αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το χάσμα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον μέσο, τους μέσους, το μέσο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χάσμα θα το καλύψει και τις σχέσεις ε, των πολιτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Άκουσα τα όσα αναφέρθηκαν στις ακροάσεις ε, και κάθε ε, επιφύλαξη που είχε εκφραστεί για την ε, ένταξη της Τουρκίας. Οποιαδήποτε επιφύλαξη αγνοήθηκε δεν ελήφθη υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεχιστεί η κατάσταση αυτών των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα μεγαλύτερη κυδαιμονική σχέση έναντι των πολιτών και σε σχέση και με τις συνθήκες της Λισαβόνας. Αυτά δεν είναι αποδεκτά. Ένα λεπτό κύριος Μπέτεν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την Επιτροπή γιατί δεν θέλω να με κατευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιασδήποτε σύσταση, αλλά υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για την καταψήφιση τούτη εδώ. Αρκετά από τα μέλη της ήταν κομμουνιστές, οι μέλη της των κομμουνιστικών κομμάτων ήταν συνδεδεμένοι με αυτά. Για παράδειγμα, ο κύριος Μπαρός, ο κύριος Σέκοβιτς, ο κύριος Φίλε, ο κύριος Πότρονικ για να αναφέρω μόνο κάποιους από αυτούς. Η κυρία Άστον ήταν ε, γραμματέας εκστρατείας κατά της, ευρωπαϊκής, ε, της πυρηνικής ενέργειας που ήταν κάτι καλύτερα από το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά κατευθυνόταν από το Σοβιετικό Μπλοκ και αυτή είναι υπεύθυνη για την εξωτερική μας πολιτική και την πολιτική άμυνας που αυτή η εξαιρετική κυρία Βαρώνη η οποία εργάστηκε για να καταστρέψει την πυρηνική ενέργεια στην ίδια τη χώρα από τη στιγμή που εμείς αντιμετωπίζαμε ε, την ε, πυρηνική απειλή. Η, η Ευρώπη γλιστρά προ την καταστροφή. Τώρα κατευθυνόμαστε από συνεργάτες των κομμουνιστών Ευχαριστούμε κύριε Μπάντεν. Ο κύριος Κέλλη και σε ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Εγώ υπερψήφισα σήμερα γιατί πιστεύω ότι από αυτές τις περιστάσεις ε, ήταν το καλύτερο πράγμα ε, να κάνει κανείς. Χρειαζόμαστε κομισιόν και τώρα έχουμε κομισιόν. Όμως θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερο σύστημα. Θα έπρεπε ένας-ένας να υπερψηφίζονται και όχι αν μπλοκ. Στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα έφτιαχνες μια ποδοσφαιριστική ομάδα, δεν θα του έφτιαχνες αν μπλοκ, αλλά θα έκρινε τον κάθε παίκτη ε, για την αξία του, για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε, να μεταρρυθμίσουμε τους ισχύοντες κανόνες, ώστε την επόμενη φορά που θα εκλέξουμε μια επιτροπή, ε, ο καθένας από του επιτρόπους θα εκλέγεται με βάση την αξία του. Αυτό θα αναγκάσει τις χώρες να προτείνουν τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους και να εξασφαλίσουν ότι θα αποδίδουν στο μέγιστο βαθμό. Θα έχουμε καλύτερη ομάδα τότε λοιπόν και μέχρι τότε προσβλέπω στη στενή συνεργασία με την Κομισιόν για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο τελευταίο συνάδελφος που θα επεξηγήσει την ψήφο του θα είναι ο κύριο Ρούμπιχ. Παρακαλώ κύριε Ρούμπιχ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που υπάρχει μεγάλη συνένεση στο Κοινοβούλιο σήμερα ζητήθηκε μια ισχυρή Ευρώπη. Η ενότητα δημιουργεί την ισχύ και γι' αυτό χαίρομαι ότι είχαμε και μια θετική ψήφο υπέρ της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι μόνο μια αποτελεσματική Ευρώπη στο τέλος τέλος μπορεί να είναι και κοινωνική Ευρώπη. Και εδώ η σαφής δήλωση και πίστη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ αυτής της θέσης είναι θετική. Αυτό μπορεί να επιμεριστεί αυτό το οποίο έχει είναι αποτέλεσμα της εργασίας μας και γι' αυτό και όσον αφορά και τις υποδομές στην Ευρώπη θα πρέπει και η έρευνα να τεθεί στο επίκεντρο και γι' αυτό είναι σχετικά απλό να κάνει κανείς τους πλούσιους φτωχούς αλλά θα είναι πιο εύκολο, πιο ευφιέσα οι φτωχοί να προσπαθήσουμε να γίνουν πλουσιότεροι και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της Ευρώπης οι φτωχοί να γίνουν πλουσιότεροι και όχι οι πλούσιοι φτωχότεροι. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Είχαμε αρκετές πολλές επεξηγήσεις ψήφου. Φτάσαμε ως το τέλος των εργασιών μας. Θα λήξει τώρα η συνεδρίαση, η ολομέλεια μέχρι τις 15.00 ε, μέχρι σε 20 λεπτά λοιπόν καλή όρεξη σε όλους σας.